Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στι ψηφοφορίε. Εγκρίνεται. Το 10 Πάμε στο σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. E l'obiezione ai sensi ε, dell'articolo 106 rinnovo della Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο στο επόμενο σημείο που έχει να κάνει με την αντίρρηση σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 106 ανανέωση έγκριση τη ενεργού ουσία μπενταζών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε για το σημείο 12. Είναι η γνωμοδότηση τζόφολη εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ε, ΔΕΔΜΗ, διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορές. Συμβιβαστική πρόταση 1, υπέρ, κατά, αποχέ ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Α, καλύπτεται. Επομένως, συμβαστική πρόταση 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπο, ε, συμβαστική πρόταση 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική πρόταση 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική πρόταση 8 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. E Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση Μπουζόη για τις ψυχοδραστικές ουσίες. Και ξεκινάμε την ε, ψηφοφορία με την τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 17 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική, που θα είναι ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. We have Έχουμε ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες. Τώρα, εάν κάποιος ε, θέλει να βγει από την αίθουσα, καλό θα είναι να το κάνει σύντομα και χωρίς φασαρία βέβαια.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 Έχουμε ανταλλαγή απόψεων τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. The στην ημερήσια διάταξη γιατί έτσι αποφάσισαν οι συντονιστές αυτό το θέμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ερίκ Τευνάγα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να μας παρουσιάσει την κατάσταση των πραγμάτων σχετικά με τις παγκότητες εγκεφαλοπάθειες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να σας παρουσιάσω την κατάσταση των πραγμάτων ε, για τον κανονισμό σχετικά με τις μεταδοτικές παγκόσμιες εγκεφαλοπάθειες. Θα είναι σχετικά σύντομη η παρουσίασή μου. Όπως γνωρίζετε, ο βασικός κανονισμός εγκρίθηκε το 2001 μεσούσεις της ε, επιζωτίας και της κρίσης ε, στη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια και τότε είχαμε ακόμα πολλά κρούσματα. Ε, ελήφθησαν λοιπόν κάποια μέτρα πάρα πολύ αυστηρά τότε. Euh, όπως θα δείτε και στις διαφάνειες, έκτοτε μειώθηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα ε, μεταδοτικών σπόγκοδων εγκεφαλοπαθειών ε, που ανοιχνεύτηκαν στην Ευρώπη. Άμα δουλεύει και η διαφάνεια θα τα δούμε κιόλας. Ωραία. Σε, μέσα σε λίγα χρόνια λοιπόν μειώθηκε κατά πολύ η εμφάνιση και ο επιπολασμός της νόσου Δύο οδικούς χάρτες εγκρίναμε έκτοτε. Τα περισσότερα από τα μέτρα της πρώτου οδικού χάρτη έγιναν κοινοτική νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την ηλικία και, και από ποια σφάγια βγάζουμε την σπονδυλική στήλη, ή ε, σε ποια υλικά επιτρέπεται να περιέχονται οστά. Ε, ε, στη συνέχεια επανήλθαν στην κυκλοφορία τα ηχθιάλευρα κτλ. Για τη δεύτερη περίοδο 2010-2015 είχαμε ένα δικό χάρτη που ήρθε να συμπληρώσει τον πρώτο. Άρα σήμερα έχουμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα σε 80 εκατομμύρια βοηθοί στην Ευρώπη είναι ελάχιστα. Πώς έχει λοιπόν σήμερα η κατάσταση. Ήδη κάποια μέτρα έχουν υιοθετηθεί και υλοποιούνται. Έχουμε αναθεώρηση τη ε, λίστα ε, υλικών ειδικού κινδύνου σε ό,τι αφορά τα έντερα των βοηδών. Ε, σταματήσαμε τους συστηματικούς ελέγχους των υγιών ζώων που σφάζονται στα περισσότερα κράτη-μέλη. την ηλικία δοκιμών για τα λεγόμενα ε, ζώα κινδύνου που είναι τα ζώα που σφάζονται εκτάκτως και πηγόντος που έχουν ψοφήσει ή που εμφανίζουν κλινικά σημεία ε, όταν εξετάζονται στο σφαγείο ακόμα ζωντανά. Επίσης, έχουμε ε, βάλει μια πιστοποίηση των κοπαδιών για τα μικρά δικαστικά την νόσο σκρέπη του προβάτου που είναι η τρομόδης νόσος του προβάτου για να βελτιωθεί ε, ε, η υγεία των ζώων. Επίσης σταματήσαμε τα ε, μέτρα εκρίζωσης για την άτυπη τρομόδη νόσο του προβάτου που δεν είναι μεταδοτική, επαναλαμβάνω όπως και η προηγούμενη. Αυτά ήταν τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει και εγκρίναμε και άλλα μέτρα εν μέρη που δεν είναι πλήρως σε εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν καθεστώς αμεληταίου κινδύνου, προσαρμόσαμε τα μέτρα αυτά για το υλικό ειδικού κινδύνου ε, και προσαρμοστήκαμε ε, στους κανόνες του ε, Διεθνούς Γραφείου Επιζωτιών. Αυτό ισχύει για τα βοηδή, για τα μικρά μερικαστικά ακόμα δεν έχει γίνει. Επίσης, ήρθε η απαγόρευση ε, ε, διατροφής ε, των μυρικαστικών με μη μυρικαστικά. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες εγγύησεις, απαγόρευση κανιβαλισμού, να μην τρώνε από το ίδιο είδος και επίσης παρακολούθηση, channeling λέγεται αυτό, της παραγωγής και με αξιόπιστους ελέγχους. Αυτό έχει γίνει για τις πρωτεΐνες που δεν προέρχονται από μυρικαστικά και προορίζονται για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Ε, δεν έχει γίνει ακόμα για τις πρωτεΐνες χείρου που προορίζονται για πουλερικά και τούμπαλι, δηλαδή πρωτεΐνες πουλερικών στη χειροτροφία. Ε, σε περίπτωση πολύ χαμηλής παρουσίας πρωτεϊνών ε, στη διατροφή θα βάλουμε ένα κατόφλι ε, αποδοχής και δράσης. Ήδη ισχύει αυτό για το μικροσκοπικό έλεγχο. Θα μπορούσε να το σκεφτεί κανείς και για άλλες μεθόδους πιο ευαίσθητες ε, στην ανείχνευση, δεν έχει γίνει ακόμα και συνεχίζουμε να προωθούμε και να ενθαρρύνουμε το γεννητικό έλεγχο για την τρομόδη νόσο του προβάτου μέσα από διάφορα προγράμματα προβατοτροφίας. Έρχομαι τώρα στα μέτρα που ε, πρόκειται να ληφθούν ή που πρέπει να ληφθούν. Αυτό αφορά τώρα τις έγιες για τη σπογκώδη και μεταδοτική εγκεφαλοπάθεια. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί ζητήθηκε η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, η οποία θα έρθει κατά το 2017 και όχι νωρίτερα, της ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια Τροφίμων. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτήσει για τη σφαγή των κοπαδιών ή των αγελών Αυτό δεν αφορά την άτυπη ε, μεταδοτική σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια των βοηδών και μόλις προσαρμόσει τους δικούς του κανόνες στο Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών θα το κάνουμε και εμείς. Αλλά αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο, πιο μακράς πνοής. Ουσιαστικά τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και τι θα κάνουμε εμείς τους επόμενους μήνες και έτη σε ό,τι αφορά την απαγόρευση ε, κάποιων ζωοτροφών, έχουμε πρωτεΐνες από έντομα τώρα. Και ο κανονισμός για τις μεταδοτικές πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες αφορά τη χρήση πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων. Ε, σήμερα απαγορεύεται η χρήση πρωτεϊνών ακόμα και από έντομα. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα να σκεφτούμε να επιτρέψουμε η πρόταση στις και στις υδατοκαλλιέργειες να χρησιμοποιούνται πρωτεΐνες από έντομα. Στη συνέχεια σε πουλερικά και μόνο αυτή τη στιγμή θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και μεθόδους εργαστηριακές αρκετά ακριβείς και αξιόπιστες θα το πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξαγωγές ε, ζωικών ε, πρωτεϊνών μυρικαστικών, σήμερα Όταν είναι κανονικά τα ζώα και καθαρά για την κατανάλωση, επιτρέπεται ε, και η εξαγωγή πρωτεϊνών, κατηγορία 3 λεγόμενη. Ε, σκεφτόμαστε να το συζητήσουμε και για τα κράτη, με τα κράτη-μέλη, συγγνώμη, προσεχώς. Αυτό αφορά μόνο τα καθαρά προϊόντα. Ενώ για τα προϊόντα που περιέχουν τέτοιου είδους υλικά, αυτό θα το δούμε σε μια δεύτερη φάση όταν θα έχουμε ε, αρκετά αξιόπιστες εργαστηριακές μεθόδους για να μπορούμε να ανοιχνεύουμε ε, ε, και να έχουμε το δίκτυο GTH που υπάρχει σε αυτά τα άλευρα και να μπορεί να ανοιχνεύεται. Και τέλος, έχουμε πρωτεΐνες για μη μυρικαστικά και χρήστη διατροφή τους. Υπάρχουν δύο δυνατότητες εκεί η χρήση ε, πρωτεϊνών από στη διατροφή των πουλερικών και το αντίστροφο, ε, πρωτεΐνες πουλερικών στη χειροτροφία. Για ε, τους χείρους είναι περίπλοκη η διατροφή τους. Στο σιτηρέσιο δηλαδή συχνά βρίσκουμε προϊόντα μυρικαστικών που επιτρέπονται όπως είναι γαλακτικές πρωτεΐνες ή ακόμα και αίμα χείρου Άρα, θα πρέπει να βρούμε μεθόδους που να μας επιτρέπουν να ανοιχνεύουμε με πάσα βεβαιότητα την πηγή των πρωτεϊνών που ανοιχνεύονται στις ζωοτροφές αυτές. Άρα, για τους Τόση ώρα μιλάω για την ε, ορνηθοτροφία, έτσι, για τα πουλερικά όπου χρησιμοποιούνται πρωτεΐνες χείρων, όχι για, την, για τη χειροτροφία. Θα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα αυτά. Ε... Συγγνώμη, λάθος τα είπα, να τα ξαναπώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο τινά να ταΐζουμε πρωτεΐνες από χείρους σε πουλερικά ή πουλερικά, ε, πουλερικών στους χείρους. Από τα πουλερικά στο χείρο σας είπα υπάρχει μια δυσκολία. Είναι περίπλοκη η διατροφή τους, είναι ε, ε, σύνθετο το σιτηρέσιο των χείρων και θα πρέπει να έχουμε μια μέθοδο εγκεκριμένη για να μπορούμε να εντοπίζουμε, να ανοιχνεύουμε. Ε, πρωτεΐνες, από ποιο ζώο προέρχονται, γιατί μπορεί να υπάρχουν πρωτεΐνες από γάλα ή από αίμα χείρου μέσα ε, στη διατροφή των πτηνών, των πουλερικών και να μας βγει ψευδός θετικό το τεστ. Θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η πηγή της πρωτεΐνης πριν εγκριθεί για την κυκλοφορία. Δηλαδή, οι πρωτεΐνες πουλερικών στη διατροφή των χείρων δεν είναι κάτι ε, το οποίο επίκειται και ούτε οι μέθοδοι PCR που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι αρκετά αξιόπιστες. Πρέπει να βρούμε πιο, πιο πιστές και πιο σύνθετες. Από την άλλη όμως, οι πρωτεΐνες χείρου που χορηγούνται στη διατροφή των πουλερικών ε, είναι κάτι το οποίο θα έρθει πιο σύντομα γιατί υπάρχουν μέθοδοι ε, που το επιτρέπουν. Και συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως που τα ε, μπέρδεψα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υλικά ειδικού κινδύνου. Euh, για τα μικρά μυρικαστικά σκεφτόμαστε να αναθεωρήσουμε τον κατάλογο και αυτό το κείμενο θα συζητηθεί στη μόνιμη επιτροπή και ε, θα βασιστεί σε γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Θυμίζω ότι σήμερα στην Ευρώπη έχουμε μόνο δύο κρούσματα ε, σφογγόδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών στα μικρά μερικαστικά και αυτό από την αρχή του 2000. Ε, δηλαδή σε εκείνη την εποχή ανάγονται αυτά. Άρα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν, το διεθνέ Γραφείο Επιζωτιών δεν προβλέπει ε, καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τα βοηθή τώρα, τα ίδια. Θα δούμε τι θα κάνει το Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών. Αναμένουμε ε, τις αποφάσεις του σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση της ε, σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών. Όπως σας είπα, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για κάποια κράτη-μέλη. Δύο κράτη-μέλη ε, δεν έχουν δει να αυξάνεται η ηλικία για τις ε, δοκιμές. Αυτά τα δύο κράτη είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Δηλαδή σήμερα θα πρέπει να κάνουν δοκιμές και σε νεαρά ζώα, υγιή, ε, τα οποία σφάζονται, φτάνουν στο σφαγείο υγιή, ηλικίας άνω των 30 μηνών και για τα ζώα που διατρέχουν κίνδυνο άνω των δύο ετών. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λοιπόν στο βαθμό που θα είναι σε θέση να μας αποδείξουν ότι μπορούν να πληρώσουν τα κριτήρια για την αναθεώρηση των προγραμμάτων παρακολούθησης θα το εξετάσουμε, αλλά δεν είναι του παρόντος. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αυτό αυτή η λεγόμενη chronic wasting disease στα αγγλικά. Είχαμε τον Απρίλιο φέτος στην Νορβηγία ένα κρούσμα. Δεν υπήρχε στην Ευρώπη αυτή η ασθένεια στο παρελθόν. Η Νορβηγία έλαβε κάποια μέτρα, πέντε κρούσματα εμφανίστηκαν σε ταράνδους ε, και σε άλλα τέτοια άγρια ζώα και λάβαμε κάποια μέτρα προφύλαξης ε, για να περιορίσουμε τις εξαγωγές από τη Νορβηγία προς τη Σουηδία και τη Φιλανδία. είναι η χρόνια εξασθενητική νόσος αυτή. Ε, κρούσματα σε άγρια ζώα, σε ταράνδους και θυράματα και ελέγχονται ε, οι εξαγωγές ε, ζώων από την Νορβήγια. Ε, θέλει προσοχή αυτή η ασθένεια γιατί δεν μεταδίδεται καθόλου ε, όπως οι άλλες πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες με, μεταδοτικές γιατί μπορεί να γίνει και μέσω του περιβάλλοντος. Και αυτή τη στιγμή γίνει αυτή η μόλυνση, είναι πολύ δύσκολο να εκριζωθεί η ασθένεια αυτή. Ε, euh, Άρα, ε, συμπέρασμα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ θετική εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ευρώπη και θα πρέπει να είναι και η απάντηση ανάλογη της ασθένειας. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές φυσικά σταδιακά και βαθμιαία και μετά από επιστημονική ε, εξέταση και αποτίμηση έχοντας όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Βεβαίως παραμένουμε σε επαφή με το διεθνή έτσι, κόσμο και αλλάζει αντίστοιχα ο κανονισμός και η νομοθεσία μας ανάλογα με το τι κάνει το Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ε, θέλω να τονίσω αυτή τη χρόνια εξασθενητική νόσο. Ε, πρέπει να προσέξουμε πολύ. Κρούσαμε και ένα να κινδυνού στην Εύσα. Τα πρώτα μέτρα ε, ε, ήθελαν να προστατεύσουν τις εισαγωγές μας και τα ζώα μας από τις αγωγές από την Ορβηγία. να δούμε τι θα πει εύσα για την νόσο αυτή. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ε, τρομόδη νόσο του προβάτου, είπαμε αυτή δεν είναι ανθρωπό ζώο νόσος, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο δηλαδή και αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία των ζώων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να διευκρινίσω τίποτα αν τυχόν χρειαστεί. Για τις πρωτεΐνες με τα ε, πουλερικά και τα γουρούνια που δεν ήταν και πολύ λαμπρή έτσι, και πεντακάθαρη η τοποθέτησή μου. Ε, παρακα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, έχετε και εσείς ξανά το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Πότση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώ γιατί υπάρχει απαγόρευση των ζωοτροφών εντόμων για τα πουλερικά, εφόσον τα, τα, τα έντομα αποτελούν φυσική τροφή για τα πουλερικά. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα. Το βασικό είναι και θα ήθελα να ρωτήσω αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει, υπάρχουν κράτη-μέλη όπου αυτές οι πρωτεΐνες πολλούνται ως ε, ε και χρησιμοποιούνται στους χείρους. Αυτό είναι γεγονός. Ε, μάλιστα και είναι αυτό που θέλει να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για κανιβαλισμό. Αυτές οι πρωτεΐνες λοιπόν πολλούνται ως λιπάσματα, μετά χρησιμοποιούνται από τους ε, γεωργούς ως ε, ζωοτροφές για τους χείρου. Το γνωρίζετε λοιπόν. Και αν έχετε λάβει γνώση, πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πεδησίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν είναι σαφές ε, από την παρουσίαση της Κομισιό ότι οι μειώσεις των περιπτώσεων ε, της ε, σπονγκόδους εγκεφαλοπάδιας μεταδοτικής ή εγκεφαλοπάδειας τα οποία έχουμε λάβει, δηλαδή η, όλη η πολιτική που ασκήσαμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει το, έχει δώσει τον καρπό της. Βρέθηκε όμως μία περίπτωση στη Γαλλία θετική και είχα κάνει ε, μία ερώτηση για, τη, για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ξέρω ότι η Κομισιό έχει ζητήσει από την ΕΦΣΑ ε, μία έκθεση για, το, για να δούμε από σε τι οφείλονται αυτά τα, αυτές οι περιπτώσεις, οι μεμονωμένες βέβαια είναι η αλήθεια. Ε, δεν ξέρω η δημοσίευση αυτή θα γίνει το 2017 ή αν υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια προκατακτικά στοιχεία. Η αν υπαρχουν καποια έχει ελέγξει τι κάνουν τα κράτη-μέλη ε, με τις ζωικές πρωτεΐνες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ζωοτροφές. Δηλαδή ποιες καταναλώνονται, ποιες χρησιμοποιούνται σαν λιπάσματα, ποιες χρησιμοποιεί, ποσοστό χρησιμοποιείται για την κομπό, κομποστοποίηση ή τι καταστρέφεται. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επομένω, μπορούμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει του κυρίου Πότσου. Είναι βεβαίω απάτη όταν χρησιμοποιούνται για αλότριου σκοπούς οι ζωοτροφές από εκείνους του οποίους προορίζονται. Τα γνωρίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται, ε, συνεργάζεται με τα κρατημέλη για να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Πάντα επαφήμεθα στις εθνικές ελεγκτικές αρχές, έτσι ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται σωστά. είναι δύσκολο να ελεγχθεί ε, μια ε, παράνομη χρήση ή απάτη, αλλά το κάνουμε παρόλα αυτά, ε, δρούμε. Σε ό,τι αφορά τα έντομα, να σας πω το εξής, προς το παρόν υπάρχει απαγόρευση η οποία ισχύει, συνδέεται με το δικό μας κανονισμό. Γιατί απαγορεύεται να χορηγείται πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης γίνεται ένα πρώτο άνοιγμα προς τις ηχθοκαλλιέργειες για λόγους κυρίως ελέγχου, να μπορούμε καλύτερα να τα ελέγχουμε για τα πουλερικά. Αυτό θα έρθει σε μια δεύτερη φάση, γιατί θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε κάθε φορά όταν βρίσκουμε πρωτεΐνες στις ζωοτροφές, να ξέρουμε ότι είναι πρωτεΐνες από έντομα. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κ. Πεντητσίνη, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ή προσανατολισμούς από την Ευρωπαϊκή, τον ε, Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, από την ΕΦΣΑ, δεν μας έχει δώσει οδηγίες. Περιμένουμε την γνωμοδότηση για το 2017. Βεβαίως, λυπηθήκαμε που εντοπίστηκε στη Γαλλία ένα τέτοιο κρούσμα, γιατί ε, από το καθεστώς αμεληταίου κινδύνου η Γαλλία πέρασε σε ένα καθεστώς ελεγχόμενου κινδύνου για μια σειρά ετών και βεβαίως περιμένουμε τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, η οποία θα έρθει περί τα τέλη του 2017, αν δεν απατώμε, για να δούμε τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα. Για τις πρωτεΐνες τώρα, δεν έχω όλα τα στοιχεία, αλλά μπορώ να επανέλθω και να σας δώσω πιο λεπτομερή έτσι, αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Όχι. Α, κύριε Γκοστέτ. Μάλιστα, θα ήθελα με βάση τα όσα είπατε, κύριε, να σχολιάσω κάτι. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Γαλλίας, λοιπόν, Είπατε εντάξει, δυστυχώς έχει αλλάξει το καθεστώς της Γαλλίας για πολλά χρόνια, όμως ξέρουμε ποια είναι η αιτία των μολύνσεων αυτών των κοπαδιών που είχαμε στη Γαλλία. Ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος, τι ακριβώς συνέβη λοιπόν. Στη Γαλλία λοιπόν ε, υπήρξε μια ενδελεχής ε, και ιδιαίτερα εμπιστευτομένη έρευνα των περιστατικών και δεν έχει εντοπιστεί η απαρχή αυτής της μόλυνσης. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει και από την ΕΦΣΑ και από τα κράτη-μέλη που είχαν ή θα μπορούσαν να έχουν τέτοια δεδομένα στη διάθεσή τους, ε, που έχουν κάνει τέτοιες μελέτες ε, τα τελευταία χρόνια, να τα διερευνήσουν για να μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτά τα φαινόμενα. Στη Γαλλία λοιπόν έχει γίνει μια εξαιρετική ε, και ιδιαίτερα επιστατωμένη ανάλυση όλων των βημάτων και δεν έχει βρεθεί το αίτιο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ για την πρωινή μας συνεδρίαση και θα ξαναλέμε το απόγευμα στις 3. Γεια σας.